Ξεκινάμε λοιπόν με τις ε, επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση GEPHAT σχετικά με την ε, εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Και θα ήθελα παρά τη φασαρία να δώσω το λόγο στον κύριο Μαστέλλα, Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες που ετέθησε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2006 ήταν να ανοίξει η αγορά και να μην υπάρχουν ε, προστατευτικοί φραγμοί, αυθαίρετα εμπόδια, ε, τα οποία οδηγούν σε διακριτική μεταχείριση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ότι η οδηγία αυτή όμω δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόσχημα για μια επικίνδυνη ρύθμιση του και με τον τρόπο αυτό να τεθούν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, το κοινωνικό dumping πλέον αντικαθίστεται από την έννοια της χώρας αποστολής και χώρας στόχο. Εγώ υπερψήφισα αυτήν την οδηγία ε, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στα κράτη-μέλη και επειδή θέλω ε, να επισημάνω τις καθυστερήσεις που υπάρχουν αλλά και κάποιες αντιφάσεις στην εφαρμογή της οδηγίας. Και σταματώ εδώ κυρία Πρόεδρε γιατί πια είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στην αίθουσα. Πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη κύριε Μαστέλα και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Μπιελάν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, ε, Αγοράς Υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θαυμάσια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με το θέμα της εφαρμογή οδηγίας για τις υπηρεσίες. Θέλουμε φυσικά ένα, μια δίκαιη ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών. Θέλουμε να διευκολύνουμε την παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ανησυχία όμως ε, διαπιστώνουμε την στάση ορισμένων χωρών που εφαρμόζουν ε, νομοθετικές διατάξεις που δεν είναι συμβατές με τις διατάξεις οδηγίας. Έτσι δημιουργούν κάποια τεχνικά εμπόδια στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 90% των νέων θέσεων εργασίας αυτή τη στιγμή δημιουργείται στην αγορά των υπηρεσιών. Γι' αυτό και η σωστή εφαρμογή της οδηγίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και νευραλγικό τμήμα της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα πρέπει ε, να προσαρμοστούν τα κράτη-μέλη στις διατάξεις αυτής της οδηγίας, προβαίνοντας η κατάλληλη νομοθετική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Grazie. La parola all'onorevole Morganti. Morganti. κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ ε, καταψήφισα την εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών, την αποκαλούμενη οδηγία Bolkenstein. Αυτή είχε ως στόχο να επιτύχει ε, συνεργασία στην Ευρώπη, να παραχθεί βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως ο στόχος τελικά της οδηγίας είναι να υφαρπαχθούν τα δικαιώματα από τις δικές μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ιταλία έχουμε τομείς αριστείας, έχουμε τα θέρετρα. Οι άνθρωποι εκεί έχουν επενδύσει, έχουν κάνει θυσίες για να αποκτήσουν μια επιχείρηση και τώρα αυτή η οδηγία θέλει να τους καταστρέψει. Ε, αυτό είναι το σύστημα, το σύστημα μιας Ευρώπης γραφειοκρατών, μεγάλων βιομηχανικών ομάδων, πολυεθνικές που θέλουν να έρθουν στην Ιταλία για να υφαρπάξουν, όπως σας είπα, τις εταιρείε μας. Εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Εμείς είμαστε με, το, με την πλευρά των μικρομεσαίων, θέλουμε να τους υπερασπιστούμε, θέλουμε να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, ε, την ε, Ιταλική υπεροχή στον τομέα αυτό. Κόσλικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ισχύουσα οδηγία για τις υπηρεσίες ζητάει από όλα τα κράτη-μέλη να άρουν τα εμπόδια και να δώσουν διευκολύνσεις στους επιχειρηματίες. Στην πράξη αυτό καθυστερεί. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η μη τήρηση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και ολιγορίες καθυστερήσεις στη δημιουργία ενιαίων θηριδών πληροφόρησης, στην ε, συνεργασία των υπηρεσιών ή την αμοιβαία ε, αναγνώριση. Πραγματικά πολύ ε, βραδία διαδικασία. Δεν δημιουργούνται ενιαίες θερίδες ενημέρωσης. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ε, για την παροχή υπηρεσιών, για τα διοικητικά, για τις διαδικασίες της κάθε χώρας, για με τρόπο εύληπτο και κατανοητό. 40% του ΕΕΠ της Ένωσης είναι υπηρεσίες. Θα πρέπει να αρθούν τα άχρηστα εμπόδια για να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες και αξιολόγησή της μας δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε σύντομα εάν αποφέρει ή όχι τους καρπούς που θέλαμε, δηλαδή την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Η εφαρμογή της οδηγίας περνάει από διάφορα στάδια. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, με τρόπο που να επιτρέπει ε, σε όλους τη νομιμότητα, τη σωστή λειτουργία. Να πρέπει να υπάρχουν σημεία επαφή σε όλα τα κράτη-μέλη, θηρίδες ενημέρωσης, έτσι ώστε να διατηρηθεί και η απαραίτητη πόρη όμως για τη λειτουργία τους. Ευχαριστώ. Grazie, la Madam Deputy Speaker, there's been κύριος Χάναν, ε, υπήρξε παρεξήγηση από την αρχή ε, της λειτουργίας Ένωσης. Τι εστί ε, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Όταν οι δική μου ψηφοφόροι ψήφισαν να μπούμε στην Ένωση και να υπάρξει η αγορά Άλλο είχαν αντιληφθεί. Δηλαδή, όταν πουλά ένα μπουκάλι νερό στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυκλοφορεί και στη Γαλλία και αλλού. Στην πράξη αυτό τι σημαίνει. Ε, τυποποίηση, ότι θα πρέπει το μεταλλικό νερό να περιέχει τα εξή μεταλλικά στοιχεία κτλ. Ο όγκος να μην είναι ε, ε, παρά μόνο μεταξύ α και β όγκου. Δηλαδή, ένα προϊόν που ποτέ δεν ε, είχε σκοπό την εξαγωγή του ε, μπορεί να απαγορευτεί στην ίδια του τη χώρα. Αυτό ισχύει και για τα αγαθά και σήμερα βλέπουμε να ισχύει και για τις υπηρεσίες. Αντί να ε, αυξάνεται η επιλογή του καταναλωτού, έχουμε μείωση περιορισμό και πολλές φορές από ένα και μόνο παραγωγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με υπερβολικές ρυθμίσεις και έτσι είναι αυτό εις βάρος του ε, ανταγωνισμού. Και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συρρυκνωθεί και στην ανταγωνιστικότητά της και η ίδια μου η χώρα. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι όταν πρωτοσυζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία η οδηγία υπηρεσιών πόσο επίμαχη ήταν και μάλιστα ήμουν εισηγητής ε, για το εμπόριο και τις υπηρεσίες και μίλησε για την ανάγκη απελευθέρωση πολλών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών, δημοσίων, ε, ταχυδρομικών, ε, ύδατος, για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να έχει μεγαλύτερο περιθώριο επιλογής ο καταναλωτής που δεν θα πρέπει να είναι έρμεο των μονοπωλίων. Και θυμάμαι τι αφιλεγόμενη ήταν τότε η οδηγία, ιδιαίτερα για τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Βέβαια, ενώ στα εμπορεύματα έχουμε μεγάλη υπηρεσία και ε, μεγάλη περιθώριο επιλογής και σε πολλές υπηρεσίες, στο ίδιο στην εκπαίδευση δεν έχουμε αντίστοιχη ελευθερία επιλογής. θυμάμαι τα κρατικά μονοπόλια παλιότερων καιρών με χαμηλή όμως ποιότητα υπηρεσιών. Θέλουμε περισσότερη απελευθέρωση των υπηρεσιών, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παντού στην Ιφίλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην επεξήγηση, σε επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Κανάν. Ε, Καντσάν πρόκειται για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Μάισνα. Που όμως, μισό λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί εμεί ε, ω φιλελεύθεροι δηλώσαμε αποχή σε αυτήν την οδηγία. Είναι πάρα πολύ καλό που έχουμε μία απόφαση. Είναι σωστό το ότι προστατεύονται οι άνθρωποι με αναπηρία. Όμω ε, αυτό ισχύει μόνο για μεγαλύτερε αποστάσει. Κατά τα άλλα, ε, πάρα πολλά που αναφέρονται δεν είναι στο ύψο τη οδηγία. Λέμε ότι αυτή η οδηγία ισχύει μόνο μετά τα 52 χιλιόμετρα. Και χώρε όπω η Κύπρο, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο λόγο εξαιρούνται, εκεί δεν υπάρχουν δικαιώματα. Αυτό ισχύει και σε άλλα κράτη-μέλη ε, που έχουν ε, γραμμές υπεραστικές ε, πάνω από 52 χιλιόμετρα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό στην Ευρώπη να έχουμε πραγματική ε, προσφορά υπηρεσιών. Τώρα λοιπόν έχουμε τους ε, επιβάτες ε, με λίγα χρήματα που δεν προστατεύονται γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποια κρατημέλη που δεν προβλέπουν δικαιώματα για τους επιβάτες και γι' αυτό δηλώσαμε αποχή. Βέβαια υπάρχουν και θετικές επιτυχέ, αλλά και αρνητικές και για το λόγο αυτό εμεί, όπως σας είπα ψηφίσαμε αποχή. Σε κύριε κυρία Πρόεδρε, η πρόταση κανονισμού ε, παρουσιάστηκε στην Επιτροπή το 2008 και τότε προβλεπόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν νέα δικαιώματα των επιβατών ε, Πούλμαν που θα μοιάζουν ε, με αυτά που έχουν επιβάτε σε άλλα μέσα μεταφορά για να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στου διάφορου διάφορους μεταφορά. Ήταν λοιπόν, είχε προηγηθεί μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και κατόπιν ακολούθησε η συνδιαλλαγή και φτάσαμε στο κείμενο επιτοπίου ψηφίσαμε σήμερα. Ένα τελικό κείμενο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πολύ καλός συμβασμός διότι εγγυάται δικαιώματα στους επιβάτες όμως χωρίς παράλληλα να επιβαρύνει τους ε, φορείς ε, που σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο βαθμό που ελήφθηκαν υπόψη τα δικά μας αιτήματα. Δηλαδή, πεδίο εφαρμογή σε δικαιώματα σε όσους διανύουν μεγάλες αποστάσεις, εξαιρέσεις ε, και τέλος ε, να υπάρχει και η δυνατότητα αποζημίωση σε περίπτωση που θυγούν τα δικαιώματα ορισμένων επιβατών. Μιλάνα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλάμε για δικαιώματα τα οποία όμω θα μπορούσαν να είναι περισσότερο εκτεταμένα. Είμαστε πεπισμένοι ότι κάτω από τα 250 χιλιόμετρα ε, τα δικαιώματα ε, των περισσότερων αδύναμων και ε, περισσότερων ηλικιωμένων δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτήν την πρόβλεψη. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ομοιογενή κριτήρια ποιότητα, όμω οι αστικέ μεταφορέ υποφέρουν πάρα πολύ στα δικαιώματα κυρίω των επιβατών. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει κανείς να προετοιμαστεί για το καλύτερο και να επαγρυπνούμε για τους μηχανισμούς εφαρμογής. Η δουλειά αυτή κρίνεται επιτυχία για το Κοινοβούλιο και είναι ένα θετικό μήνυμα ε, προς όφελος των ε, πολιτών. Όμως ο συμβιβασμός ε, αφορά πάντα τη μέση οδό, ε, κατ' ουσίαν εμείς ε, δείξαμε ότι είμαστε καλοί αναγνώστες ε, των, των αναγκών, όμως το Συμβούλιο από την άλλη πλευρά δυστυχώς εκφράζει άλλα συμφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ούτζας. Grazie Presidente. Io vorrei complimentarmi con l'onorevole Cancian per il lavoro. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καντσάν για την πολύ καλή δουλειά που έκανε στο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ε, δεν συμφωνώ όμως με τον κύριο Μαστέλα που λέει ότι αυτό, αυτή η διάταξη και αυτή η ρύθμιση είναι μεγάλο επίτευγμα για τους πολίτες. Γιατί αυτοί προστατεύονται μόνο εφόσον κάνουν μια διαδρομή πάνω από 250 χιλιόμετρα. Πού είναι όμως η προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών πολιτών. Όπως είπε, ε, είπαν και οι προηγούμενοι συνάλφοι, Ολόκληρες χώρες, η Κύπρος, ε, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, εξαιρούνται από αυτή τη ρύθμιση. Γι' αυτό λοιπόν η δική μας ομάδα ψήφισε αποχή. Δεν καταψηφίσαμε γιατί υπάρχουν και κάποια δικαιώματα που προστατεύονται και ως ε, εκ τούτου ε, θεωρώ ότι πράγματι προστατεύονται σε κάποιο βαθμό τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γι' αυτό δηλώσαμε αποχή. Κατά τα άλλα όμως θέλω να σας πω ότι πρέπει να μεριμνήσουμε ταχύτητα έτσι ώστε να, πράγματι να προστατεύσουμε επί της ουσίας τα δικαιώματα των επιβατών. Επόμενος ομιλητής παρακαλώ, επόμενος ε, αγορητής, ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε και να μεριμνήσουμε για τα δικαιώματα των πολιτών. Όταν όμως μιλάμε για δικαιώματα θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τις υποχρεώσεις. Δεν νοούνται δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις και ευθύνες. Όταν εξετάζουμε την πρόταση αυτή για την προάσπιση των δικαιωμάτων των επιβατών ε, λεωφορείων και πούλμαν, διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ θετική. Βλέπουμε όμως ε, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, υπάρχουν ε, πολύ μικρές εταιρείε, οικογενειακές και διαρωτόμαστε αν είναι σκόπιμο να επιρρύπτουμε τέτοιο βάρος και να αυξάνουμε το άχθος για τις οικογενειακές αυτές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλά αντικρώμενα μερικές φορές συμφέροντα. Η προστιθέμενη αξία της πρότασης αυτής έγκυται στην προστασία των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα και χαίρομαι που ελήφθησαν οι δικές τους ανάγκες υπόψη ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ταξιδιού για αυτούς. Η πρόταση πάντως είναι κάπως επίμαχη γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για δικαιώματα ξεχνώντας τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες. Θα πρέπει επίσης να μην είναι δυσανάλογο ε, το κόστος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα τον κανονισμό αυτό. Ακόμα και αν θεωρώ ότι σίγουρα δεν πήγαινε αρκετά μακριά. Είναι μια αρχή, εν περιπτώσει, και κάποια στιγμή στο Κοινοβούλιο και ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε βρεφικά βηματάκια, αλλά δεν πειράζει. Κάποια κράτη-μέλη ε, είναι εκτός του κανονισμού, βεβαίως, ε, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες από 250 χιλιόμετρα. Και εγώ θα προτιμούσα τη γραμμή των φιλελευθέρων που ζητούσαν πολύ μικρότερες αποστάσεις και διάρκεια ταξιδιού. Εν πάση περιπτώσει, μερικά από τα βασικά δικαιώματα του κανονισμού ε, αφορούν ταξιδιώτες και επιβάτες σε μικρότερες αποστάσεις και αυτά είναι άτομα με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα. Και ε, να μην υπάρχει δηλαδή ε, διάκριση στην πρόσβαση και να είναι καταρτισμένο το προσωπικό για οι εργαζόμενοι για τα θέματα αυτά. Αλλά η περίοδος ε, παρέκκλησης και εξέλιξης ε, είναι μέχρι μια δεκαετία. Ε, ξέρω ότι οι εταιρείε χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη το συντομότερο και του ζητώ να εφαρμόσουν αυτό το κανονισμό. Ευχαριστούμε πολύ. το λόγο έχει ο κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, εγώ είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των επιβατών ε, στα λεωφορεία και πούλμαν και υπέρ τη ενίσχυση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα. Αλλά δεν με ικανοποιεί πλήρω η συμβαστική λύση. Επίση, το όριο των 200 χιλιόμετρων θα ε, επέτρεπε στην Ιρλανδία να αποκλείσει της ε, την Ήπεθρο, το, τη Δυτική Ντόνεγκαλ, Γκόλγουεϊ κτλ γιατί οι περισσότερες περιοχές βρίσκονται εκτός των 250 χιλιόμετρων. Επίσης, το δικαίωμα αποζημίωσης, σε παραλαμβάνω, φέρνει σε δυσμενή θέση αυτούς που διαμένουν στην Ήπεθρο σε μικρές χώρες. Και το κόστος ασφάλειας είναι απαγορευτικό και θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλές εταιρείε. Δεν υπάρχουν εναλλακτικέ άλλωστε συγκοινωνίες σε, περιπτώσεις αυτές. Βέβαια θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση που λάβαμε σήμερα, αλλά η περίοδος ε, εξαίρεσης θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία σε αυτούς που βρίσκονται πέραν των 250 χιλιόμετρων να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Επί της αρχής συμφωνώ και επί της ουσίας, αλλά για τους προαναφερθέντες λόγους χρειάστηκε να κρατήσω στάση εποχής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πάνω από 70 εκατομμύρια πολίτες στην Ένωση χρησιμοποιούν καθημερινά λεωφορεία. Γι' αυτό έχει έρθει η ώρα να ισχύσει ένας κανονισμός που να ε, προστατεύει τους επιβάτες αντίστοιχα με τους επιβάτες των αεροπλάνων ή των τρένων. Ανεξάρτητα από την απόσταση έχουν 12 θεμελιώδη βασικά δικαιώματα επιβάτες. Στη συνέχεια έχουμε αυτό το θέμα των 250 χιλιόμετρων που έχουν ε, το δικαίωμα αξίωσης αποζημιώσεων σε περίπτωση καθυστερήσεων ή απώλειας αποσκευών. Για τα μικρότερα κράτη, ωστόσο, αυτό το όριο των 250 χιλιόμετρων απόσταση είναι παράδεκτο. Επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια σε άτομα με αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα όπως ισχύει στις αερομεταφορές. Στο μέλλον θα υποστηρίξω ένα κοινό κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών όλων των μέσων μεταφοράς. Και αυτό θα είναι πιο απλό και για τους χρήστες. Ευχαριστώ. Μικολάζικ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα δικαιώματα των επιβατών ε, λεωφορείων και πούλμαν ε, θα πρέπει να είναι σαφώς ρυθμισμένα στην Ευρώπη. Όπως ισχύει για τις αερομεταφορές και το σιδηρόδρομο. Θεωρώ καλό συμβιβασμό το σημερινό κείμενο του κανονισμού. Χαίρομαι που ρυθμίζονται σωστά πλέον τα δικαιώματα των επιβατών και θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα. Επίσης το θέμα των ε, αποζημιώσεων για ε, θέματα ατόμων με αναπηρία πάλι για τα αναπηρικά αμαξίδια ή ακόμη και η κατάρτιση του προσωπικού ε, για θέματα αναπηρίας. Είναι πολύ καλά και θετικά και κατά των διακρίσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση διότι είναι σαφέστατα βελτίωση της σημερινής κατάστασης. Ισορροπημένη ήταν η λύση τελικά που προστατεύει και τα δικαιώματα των επιβατών αλλά δεν απειλεί, ε, μάλλον εξασφαλίζει την ύπαρξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 250 χιλιόμετρα είναι το πεδίο εφαρμογή και τώρα έχουν δικαίωμα οι επιβάτες σε περίπτωση ακύρωσης, overbooking ή καθυστέρησης άνω των δύο ώρων. Ε, Πολλέ φορέ οι εταιρείε αυτές είναι μικρομεσαίες ε, που μπορεί ε, η υποχρέωση αποζημίωση να του φέρει στα όρια της επιβίωσης. Καλή είναι λοιπόν η λύση για να μην είναι άπειρη η αποζημίωση. Και χαίρομαι για τα 250 χιλιόμετρα. Δεν απαγορεύεται ποτέ να έρθει μια νέα νομοθεσία κάποια στιγμή αν χρειαστεί ενδεχομένω κάτι πλέον να βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Κάντσιαν, τον εισηγητή. Η σημερινή έκθεση, η έκθεση που ψηφίσαμε είναι καλός συμβιβασμός, διότι προστατεύει έτσι τα δικαιώματα των επιβατών ώστε να μην ε, υπάρχει κίνδυνος για τις εταιρείες ε, το λεωφορείο που είναι μικρομεσές. Βελτιώνονται επίσης και οι προϋποθέσεις και τα δικαιώματα των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα. Ε, όλα αυτά θα βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Καντσάν για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε και κυρίως ε, για το αίσιο αποτέλεσμα της ε, συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο. Ο συμβιβασμό ε, κάτω από το πρίσμα της εφαρμογής αφορά στο ότι στην πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνονται 12 σημαντικά δικαιώματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ε, προστασίας ε, των δικαιωμάτων, κυρίως ε, των ατόμων με αναπηρία και θα ήθελα να αναφερθώ πάνω απ' όλα στο ότι δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση, να προβλέπονται οι απαραίτητοι εξεπλισμοί να ενημερώνεται το προσωπικό των πούλμαν και των λεωφορείων για την αναπηρία. Αυτέ οι πληροφορίε πρέπει να δίνουν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό που ενδιαφέρει επίση είναι να προστατεύουμε τα δικαιώματα, χωρί όμω να επιβαρύνουμε του μεταφορεί. Ε, γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει και δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε ένα τεράστιο βάρο που θα είχαν να αντιμετωπίσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Ντότ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αναγνωρίζω τα πολυάριθμα θετικά στοιχεία της έκθεσης αυτής και είμαι αναφαδόν υπέρ του δικαιώματος των αναπήρων να έχουν πρόσβαση στις μεταφορές και στο δικαίωμα αποζημίωσης. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι τέτοιου είδους συστήματα και διατάξεις θα πρέπει να θεσπίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και το οικονομικό κόστος που συνοδεύει την πρόταση θα είναι απαγορευτικό για πολλούς παρόχους ε, υπηρεσιών μεταφορών. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι πολλές τέτοιες εταιρείες ε, λεωφορείων και πούλμαν είναι ιδιωτικές, πολλές φορές οικογενειακές και υφίστανται τεράστια οικονομική πίεση εξαιτία της ε, ε, των τιμών ε, καυσαερίων τους τελευταίους 18 μήνες. Με τέτοιες προτάσεις για αποζημίωση το μόνο αποτέλεσμα θα είναι οι υψηλότερες τιμές ναύλων και εισιτηρίων για τους ε, επιβάτες και απειλή για κλείσιμο πολλών ε, εταιριών. Νομίζω ότι υπάρχουν και αρνητικέ πτυχές σε αυτή την ε, απόφαση. Ο κύριος Φιντάντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ήταν μια μεγάλη διαδρομή αυτή που τελικά μας οδήγησε σήμερα στο να ψηφίσουμε για αυτήν την έκθεση. Και θα ήθελα μαζί με τους άλλους ανθρώπους, να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Καντσάν, ο οποίος αυτή την ε, διαδρομή την διένυσε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα λοιπόν υπάρχει ένας πολύ σωστός κανονισμός όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών και νομίζω το επόμενο βήμα είναι να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο κείμενο ε, το οποίο θα ενώνει όλες αυτές τις σε ένα και μόνο κείμενο. Ε, πράγμα, το πεδίο εφαρμογή είναι πολύ λογικό. Το θέμα όμω ε, είναι να συμπεριλάβουμε όλε τι χώρε. Γιατί τώρα ξέρονται βία. Καλό και αυτό. Πάρα πολλά, πάρα πολλά άρθρα είναι υποχρεωτικά ε, μετά από 250 χιλιόμετρα. Ε, άκουσα σήμερα το πρωί να αναφέρεται από ορισμένου συναδέλφου στη συζήτηση κάτι το οποίο μέχρι τώρα πολλοί διέψευσαν. Δηλαδή είπαν ότι πρόκειται για μεγάλη προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για ένα συμβιβασμό ε, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Πριν δώσω το λόγο ε, στον συνάδελφο κύριο Όβιρ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ε, να αναφέρω ότι για να ζητήσει κανείς το λόγο κατά τη διάρκεια των επεξηγήσεων ψήφου θα πρέπει να το έχει ζητήσει γραπτά ημέρες πριν από την δυνατότητα που του προσφέρεται να προβεί σε επεξήγηση ψήφου. Η κυρία Όβιρ. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε που δεν είχα υποβάλει εμπρόθεσμα το αίτημά μου για επεξηγήση ψήφου. Ψήφισα κατά τη έκθεση αυτής γιατί δεν εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των επιβατών σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς. Η έκθεση αυτή άλλωστε δεν καλύπτει τα μικρά κράτη-μέλη. Στην περίπτωση των μικρών κρατών μελών, η οδηγία αυτή θα εφαρμοστεί μόνο μερικώς. Οι επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν είναι κυρίως νέοι και όχι ιδιαίτερα εύποροι. Γι' αυτό και ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής και της πρότασης. Ευχαριστώ. Περάμε τώρα στις ε, επεξηγήσεις ψήφου της έκθεσης Κάλαναν για τις προδιαγραφές απόδοση όσον αφορά τι εκπομπέ καυσαερίων από καινούργια ελαφρά εμπορικά οχήματα. Δίνω πρώτο το λόγο στον κύριο Γκζιμπ. Ευχαριστώ. Καταλήξαμε στη συμβαστική λύση για το θέμα αυτό τις εκπομπές καυσαερίων σε ελαφρά εμπορικά οχήματα μεταξύ των Επιτροπών Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε να μειώσουμε στα, ε, στα επίπεδα από 230 σε 140 σε, μέσα σε 10 χρόνια. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση για το κόστος των χρηστών σε ό,τι αφορά ε, και την αύξηση των τιμών αυτών των ε, εμπορικών οχημάτων. Βέβαια, κυρίως οι εταιρείες αυτές είναι μικρές, οικογενειακές και σκεφτήκαμε κάποια δυνατότητα υποστήριξης ε, χρηματοοικονομικής ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Ένωση προς μικρές αυτές επιχειρήσεις. Γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε κάποια φράγματα στην ανάπτυξη αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ελπίζω να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να μην γίνει αυτή η πρόταση για, για τον περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και, ευχαριστώ να... και ελπίζω να εφαρμοστεί λογικά αυτός ο κανονισμός. Το λόγο έχει ο κύριος Γιάρ. Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ε, ένα μακροπρόθεσμο φιλόδοξο πάγιο στόχο που κατάφερε να τον επιβάλλει απέναντι στα άλλα όργανα. Τα 147 ε, γραμμάρια ένα χιλιόμετρο τελικά καταλήξαμε με καινοτομία ε, όμως και τεχνολογία θα επιβληθεί αυτός ο στόχος. Είναι πιο καθαρά τα αυτοκίνητα, αλλά ε, παραμένουν ταυτόχρονα προσιτά για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες χρήστες. Ε, γιατί δεν βοηθάει ούτε το κλίμα να είναι πανάκριβα τα νέα καθαρά αυτοκίνητα και να συνεχίζουν να ρηπαίνουν οι επαγγελματίες γιατί δεν μπορούν να τα αγοράσουν και χρησιμοποιούν τα παλιά τους. Χαίρομαι λοιπόν για το αποτέλεσμα και που εγκρίθηκε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Η κυρία Φόρντ με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ψηφίσαμε τώρα για αυτά τα ελαφρά οχήματα και ε, έχουμε πάλι ένα μεγάλο επιβλητικό τίτλο ε, για κάτι το πολύ απλό. Εδώ μιλάμε κυρίως για μικρά φορτηγά ε, και τα επίπεδα απόδοση ε, κατ' ουσίαν μιλάει, αναφέρεται και εννοεί τις εκπομπές διοξιδίου. Οι κατασκευαστές και οι απλοί βιοτέχνες που έχουν το δικό τους το φορτηγάκι. Είναι ζωτική σημασία το φορτηγάκι αυτό για αυτούς ε, και ε, οι εκπομπές διοξιδίων πάντα ήταν βέβαια ένα καθοριστικό ε, στοιχείο. Τώρα όσον αφορά τη δική μου εκλογική περιφέρεια στη γραμμή παραγωγής έχω δει να υπάρχουν κάποιες καινοτομίες που προέρχονται από την ίδια την εταιρεία. Ορισμένοι πιστεύουν ότι επειδή εδώ ορίζονται κάποιοι στόχοι ότι και αυτοί θα επιτευχθούν. Όμως η αλήθεια είναι ότι το να επιτύχει κανείς αυτό αυτούς τους ε, στόχους ε, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει καινοτομία είτε για τα φορτηγάκια είτε για οτιδήποτε άλλο και αυτό προκύπτει μετά από ε, ζήτηση από τους καταναλωτές και δεν προέρχεται απλά και μόνο από την θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας. Ευχαριστούμε πολύ. Κέλλη παρακαλώ. Δυστυχώς ε, δεν ε, ήμουν παρόν στη συζήτηση γιατί συνέπιπτε με μια άλλη συνεδρίαση που είχα. Γι' αυτό σας ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε το λόγο να πω δύο λόγια τώρα. Η στρατηγική του 2020 με τους φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό όμως να υλοποιήσουμε τους στόχους και για την ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα για τα εμπορικά οχήματα και τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Τα εμπορικά οχήματα βρίσκονται στον δρόμο κάθε μέρα και διανύουν τεράστιες αποστάσεις. Με μια τέτοια οδηγία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020 για την αποτελεσματικότητα του καυσαέριου, γιατί κάτι τέτοιο θα εξανάγκαζε τους κατασκευαστές να τροποποιήσουν τους κινητήρες για να γίνουν πιο αποδοτικοί και το κόστος ε, θα ήταν ε, τεράστιο για τους αγοραστές ε, ενώ το περιβαλλοντικό κόστος επίσης θα ήταν πολύ μεγάλο. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου για την σύσταση, λένε, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ε, και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαστέλα. Παρακαλώ κύριε Μαστέλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, το Συμβούλιο μας έστειλε την πρόταση για απόφαση που εξισιοδοτεί την διαδικασία της ενισχυσμένης συνεργασίας για να υπάρχει ένα ενιαίο δίπλωμα ευρυστεχνίας και αυτό αφορά ορισμένε χώρες. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι κατά αυτού του συστήματος. Πρόκειται για ένα σύστημα τρίγλωσσο που τελικά θα κατέληγε σε διακριτική μεταχείριση και αποτελεί κατάφορη παραβίωση της ισότητας και ισοτιμίας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα λοιπόν ε, θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να εγκριθεί αυτή, αυτός ο κανονισμός και για νομοθετικούς και άλλους θεσμικούς λόγους ε, θα έπρεπε να περιμένουμε και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες και αυτή θα ε, διαλευκάνει όχι μόνο τεχνική φύσεως θέματα αλλά πάνω απ' όλα και τις ε, νομικές συνέπειες. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος δρόμος και γι' αυτό το λόγο εγώ καταψήφισα. Πολύ ωραία. Ρόντε παρακαλώ. Ο κύριος Ρόντε. Η συζήτηση έγινε στο Κοινοβούλιο για την ενισχυμένη πλειοψηφία, ενισχυμένη συνεργασία ε, όσον αφορά το ε, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Ε, δεν αρκεί εδώ να χαμογελάει κανείς. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολιτικοί που λένε ότι το σημαντικότερο θέμα είναι η διαφύλαξη της γλώσσας τους και τώρα λένε ότι παρόλα αυτά επιθυμούν να συνεργαστούν. Μα είναι παράδοξο. Σήμερα δεν υπάρχει κοινή αγορά αυτό το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνία ε, θα κοστίζει 10 ε, φορές παραπάνω από ότι το να το αποκτήσει ε, κανείς στι Ηνωμένε Πολιτείε. 250 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το επιπρόσθετο κόστος. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να καταψηφιστεί η ενισχυμένη συνεργασία και ορισμένες χώρες να πάψουν να ε, δημιουργούν τροχοπέδι, να προκαλούν τροχοπέδι και φραγμούς αυτή τη ε, διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπιέλαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και 20 χρόνια στο, σε Ευρωπαϊκό Φόρα συζητούμε αυτό το θέμα της ε, ενιαίας προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα και ε, το Αμερικανικό σύστημα πιστοποίησης και καταχώρησης δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ επιβαρυντικό. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουμε την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη γιατί με τον ραγδαίο παγκόσμιο ανταγωνισμό δεν μπορούμε να αποφεύγουμε τη λήψη αποφάσεων για τέτοια θέματα. Χρειαζόμαστε ενισχυμένη λοιπόν συνεργασία για την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε και διάφορα επίμαχα ζητήματα όπω το γλωσσικό. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος μικρότερων, λιγότερο πυκνοκατοικημένων και συνήθως και λιγότερο οικονομικά εύπορων χωρών. Ευχαριστώ. Παρόλα l'onorevole Παλώνε. Παλώνε παρακαλώ. Κύριος ε, ζούμε σε μια εποχή όπου ε, οι επιχειρήσεις μας είναι ε, εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό τα, διπλωματικά, τα διπλώματα αυτά ευρεστεχνίας ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ως στόχο να περιορίσουν ε, το κόστος για να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Και διαρωτώ με, δεν θα ήταν καλύτερα ε, να έχουμε δίπλωμα ευρεστεχνίας μόνο σε μία γλώσσα και έτσι να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζουμε όλοι, στην Ευρώπη έχουμε δύο νομικά καθεστώτα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω λοιπόν Λοιπόν, θα ήταν περισσότερο σκόπιμο να εναρμονίσουμε αυτά τα νομικά συστήματα. Και τέλος, το να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία, αυτό όχι μόνο αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά είναι και ένα εμπόδιο ε, το οποίο δημιουργεί στρέβλωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, γιατί προφανώς ε, θα υπάρξουν κράτη-μέλη τα οποία θα είναι λιγότερο ευνοημένα από άλλα. Πολύ ωραία. Μπυρίλο, παρακαλώ. Επόμενος αγωνιτής, ο κύριος Μπυρίλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ο στόχος ε, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολλά χρόνια να επιτύχουμε ένα σημαντικό εργαλείο που είναι το ε, κοινοτικό δίπλωμα ευρωσιτεχνίας που θα επιτρέψει επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ανταγωνιστεί με τα ίδια όπλα. Ε, είμαστε όμως αναγκασμένοι να διαπιστώσουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα ε, ζημιώνει παραδείγματος χάνει την ε, Ιταλία. Η απόφαση να υπάρχει το δίπλωμα αριστεχνίας μόνο σε τρεις γλώσσες. Αυτό θα προκαλέσει ανισότητα, ε, θα ζημιώσει τις ιταλικές επιχειρήσεις ε, κυρίως ε, που δεν θα καλύπτονται από το προτινόμενο γλωσσικό καθεστές. Πριν από κάποιους μήνες εγώ κατέθεσα στην Επιτροπή μια εξαίρεση για να προστατεύσω τη χρήση της ιταλικής γλώσσας. Βλέπω όμως ότι τώρα υπάρχουν και άλλες χώρες που θα ζημιωθούν και για όλους αυτούς τους λόγους εγώ οδηγήθηκα στην αποχή. Το λόγο έχει ο κύριος Γκζίμπ. <clears throat> Ευχαριστώ. Οι προτινόμενες διατάξεις για την ε, προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνία ε, είναι σημαντικέ. Οι μέχρι τώρα διατάξει δεν ικανοποιούσαν κανέναν. Η ενιαία προστασία είναι σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη και των χωρών μεμονωμένα, αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα στηρίξουμε την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Μία ενιαία προστασία με ένα πλούστερο σύστημα ε, περιέχει και κάποια επίμαχα σημεία όπως ε, την αναφορά μόνο σε τρεις γλώσσες, αλλά υπήρχε κάποια πρόοδο σχέση με τις προηγούμενες προτάσεις. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν ε, το οικονομικό, την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την προστασία των διπλωμάτων ευρωστηχνίας. Επίσης, ε, έχουμε και το νέο όρο του Sleeping ε, Innovators. Το αναφέρουμε αυτό στην Επιτροπή Βιομηχανίας, αυτέ αυτού είδου της βιομηχανίας θα πρέπει να τις αθαρρύνουμε να δώσουμε ενάυσματα για καινοτομία, αλλά και για κατοχήρωση με διπλώματα βριστεχνίας των ε, εφευρέσεών τους. Οι νέες ε, νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να προστατεύσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και να κατοχυρώσει τα διπλώματα ευρεσιτεχνία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Grazie, la parola ora all'onorevole Le Grip, prego. Λεγκρίπ παρακαλώ. Η κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση Λένε που δίνει την άδεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενισχυμένη συνεργασία έτσι ώστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ένα ενιαίο δίπλωμα ευαισθητεχνίας. Επιτέλους θα έλεγα 20 χρόνια αγώνων για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα μια πρώτη απόπειρα διπλώματος, ε, κάτι που περιμένουν εδώ και χρόνια οι εταιρείε μας. Είναι μείζον ε, μέσω ενίσχυσης της ε, ανταγωνιστικότητάς τους. Δίνοντας αυτή την άδεια, την έγκριση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δείχνει πόσο ενδιαφέρεται για αυτή την ιδιαίτερη μορφή ενισχυμένη συνεργασία. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη μόνο φορά που εφαρμόζεται. Ε, στέλνει όμως ταυτόχρονα ένα πολύ θετικό και συγκεκριμένο μήνυμα για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Ακούσαμε ότι 25 από τα 27 κράτη-μέλη εντάσσονται στην ισχυμένη αυτή συνεργασία για τη δημιουργία νέου διπλώματος τεχνίας. Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν γνωρίζω ε, μάλλον τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν στα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα, στο κάνουμε επιτέλους. Είναι πολύ σημαντικό και για τη βιομηχανία μας. Η κυρία Πιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απήχα εγώ στην ψηφοφορία γιατί θεωρώ η απόφαση δημιουργία νέου διπλώματο ευρεσιτεχνία με την ενισχυμένη συνεργασία είναι ακόμα μία αποτυχία του Συμβουλίου. Μόνο 9 κράτη-μέλη συμφώνησαν και αναγνωρίζει και το ίδιο το έγγραφο ότι δεν προλαβαίνουν αυτά φτάσουν στου στόχου του ε, εγκαίρω σε λογική ε, διάρκεια. Επίσης ε, υπάρχει και το θέμα το γλωσσικό. Θα έπρεπε το Συμβούλιο να είχε καταβάλει προσπάθεια να καταλήξει κοινή θέση και ενδεχομένως να εργαστεί περισσότερο ε, για τη χρήση μίας και μοναδικής γλώσσας. Λαμβάνοντα ε, υπόψη πόσες γλώσσες έχουμε και πόσα μητρώα καταχώρησης. Χρειάζεται μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και πάλι μια εθνική αντίληψη των κρατών μελών μας οδήγησε εδώ τρεις γλώσσες μόνο. Με τέτοιου είδους μέτρα δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχουμε την εδραίωση και την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού μοντέλου. Σας ευχαριστώ. Μικολάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνουμε πρώτοι παγκοσμίω, θα πρέπει να αξιοποιούμε την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά εμπόδια για την ε, ενιαία ευρεσιτεχνία και την ανάπτυξη περαιτέρω της ενιαίας αγοράς. Αυτό που θα ρίνει τους εφευρέτες στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση της ε, διαδικασία αυτή με ενιαίο ε, δίπλωμα και ενιαίο δίκαιο τεχνίας. Έτσι θα μπορούν να έχουν καλύτερη επισκόπηση της κατάστασης οι εταιρείε και οι μικρομεσαίες, γιατί για αυτούς το κόστος είναι υψηλότερο από ότι σε αντίστοιχε εταιρείε των ΗΠΑ. Γίνονται προσπάθειες λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή για μια ενιαία προστασία με ενιαίο δίπλωμα τεχνίας. Μέχρι σήμερα όμως αυτή η προσπάθεια είχε να βαγίσει. Γι' αυτό πιστεύω πλέον ότι πρέπει να υπερψηφίσει αυτή την προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πριν από ένα αιώνα, όταν δεν αναγνωριζόταν ε, το δίπλωμα τεχνίας από την αμερικανική ε, τηλεφωνία, αυτό δεν ήταν επειδή δεν ήταν στα αγγλικά ή στα ιταλικά, αλλά γιατί δεν κάλυπτε τις προδιαγραφές. Δεν υπήρχαν τα χρήματα για να καταγραφεί αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και πέρα από την ψήφο ή τη σημερινή ψηφορία, εγώ θεωρώ το γεγονός ότι θα μπορούσε να υπάρχει ε, ένα τρίγλωσο κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνία χωρί τα Ιταλικά, αυτό είναι προφανώ ε, αδυναμία τη δική μα κυβέρνηση. Δηλαδή δεν μπορεί να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό αποδεικνύει την αδυναμία τη δική μα πολιτική. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην καινοτομία και στην έρευνα και θέλω να επενθυμίσω ότι η μελέτη για την ανταγωνιστικότητα που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβρη αναφέρει πω η Ιταλία τα τελευταία χρόνια χάρισε με άνεση 4 ε, δις ευρώ σε άλλες χώρες ε, που έχουν ερευνητές. Ε, η χρήση λοιπόν της Ιταλικής γλώσσας από ό,τι φαίνεται δεν εξυπηρετεί πια γιατί όλοι θα μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά για να μπορούν να παρουσιάζουν τα δικά τους τα διπλώματα ευρυσεχνίας στην Ιταλία. Αντινόρο παρακαλώ, κύριος Αντινόρο. Ευχαριστώ πρόεδρε εγώ ε, λαμβάνω το λόγο ε, για να εξηγήσω γιατί καταψήφισα σήμερα ε, διότι αυτή η δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα μπορούσε να ωφελεί στην Ευρώπη αλλά στη τελική ανάλυση το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ καλύτερο εάν είχαμε ακολουθήσει μια διαφορετική διαδικασία. Δηλαδή ε, με αυτή την ενισχυμένη συνεργασία δεν οδηγούμεθα πουθενά. Αυτό είναι απλά μια νέα φάση στην μακρά ιστορία ε, κοινωτικού διπλώματος που ξεκίνησε ήδη τη δεκαετία του 1990. Εγώ λοιπόν ε, καταψήφισα αυτό το ψήφισμα γιατί είναι ασυμβίβαστο με αυτά που προβλέπει το άρθρο 20 της συνθήκης. Η πρόταση της ε, Επιτροπής ε, δεν αφορά το σύνολο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 118 και στη τελική ανάλυση θεωρώ ότι θα παρεμποδίσει την ελεύθερη μετακίνηση, διακίνηση κεφαλαίων. Από πλευράς πολιτικής θα ήταν πολύ πιο κομψό και πολύ πιο σωστό να περιμένουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ε, θα εκδοθεί στις 8 Μαρτίου. Τώρα ε, νομίζω ότι θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να αναθεωρήσουμε τη θέση μας. Σας όλοι παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά είδαμε την ανικανότητα της Ιταλικής κυβέρνησης να προστατεύσει το ευρωπαϊκό προφίλ ε, της Ιταλίας, να προστατεύσει τα συμφέροντα της ε, βιομηχανίας μας. 25 χώρες από τις 27 και η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνούν σε μια πρόταση που ρυθμίζει τα θέματα των διπλωμάτων ευρωστεχνίας ε, κυρίως βοηθούν τις καινοτόμες υπηρεσίες. Αποκλείεται λοιπόν η Ιταλική βιομηχανία, αυτό θα επιβαρύνει τις δικές μας ε, τις επιχειρήσεις, δεν θα προστατεύονται επαρκώς ούτε στην Ευρώπη ούτε σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια κυβέρνηση λοιπόν που δεν κάνει τίποτα για να διαδώσει τον Ιταλικό πολιτισμό στον ε, κόσμο, ε, δεν εκμεταλλεύεται την Ιταλική γλώσσα, μια χώρα που έχει όμως το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη πολιτιστική κληρονομιά του κόσμου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 λύνεται το θέμα το γλωσσικό με σοβινιστικό τρόπο. Ενώ οι δικές μας επιχειρήσεις ζήτησαν τελικά τα διπλώματα να είναι μόνο στα αγγλικά, γιατί αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί η παγκόσμια οικονομία. Το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι ότι δεν μπορεί κανείς ε, να καταθέσει τα διπλώματα που στη δική του τη γλώσσα. Ο συνάδελφος κ. Μπαρνιέ ζήτησε ε, ταχύτατα να ε, ψηφιστεί το θέμα πριν όμως από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που όπως ξέρουμε ε, θα εκδοθεί την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Θα είναι μια απόφαση που θα αφορά κυρίως σε δύο θέματα. Πρώτον στη χρήση της εθνικής γλώσσας για να ε, μπορεί κανείς ε, να προστατευτεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεύτερον την νομιμότητα των δικαστηρίων να αποφασίζουν για τα διπλώματα ευρωστεχνία. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να περιμένουμε πριν προχωρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν η δική μα απόφαση, η απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματο και τη Ιταλική Αντιπροσωπεία είναι να δηλώσουμε αποχή. Πολύ ωραία. Επόμενο αγορητή, ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ. Σίγουρα η πρόταση αυτή δεν είναι τέλεια και μάλλον θα πρέπει να επανεξεταστεί μετά την ε, αναμενόμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που την περιμένουμε σε λίγες εβδομάδες. Φυσικά όμως είναι και ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση και αυτό και την υποστήριξα. Παρακολούθησα πολλά και διάφορα σεμινάρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα την καινοτομία. Η General Electric ε, ε, πραγματοποίησε κάποιες δημοσκοπήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι η πρόοδος μετά από μια ύφεση θα πραγματοποιηθεί μόνο χάρη στην καινοτομία, που σημαίνει έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και νέα προϊόντα. Τα νέα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτονται από ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Και όσο πιο εύκολο αυτό, τόσο καλύτερο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι εύκολο και ε, με σωστή αναλογία κόστου ωφέλου, αντίστοιχο και εφάμιλο με το αμερικανικό. Αυτό είναι ο απότερο στόχο. Αυτό είναι ίσω το πρώτο βήμα. Γι' αυτό και τάχθηκα υπέρ της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αποχή ψήφισα εγώ. Στην έκθεση λένε όχι γιατί έχω κανένα πρόβλημα με τη δημιουργία του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το αντίθετο, οι επιχειρήσεις στη Φλάνδρα το ζητούν εδώ και καιρό την ίδια την ιδέα δεν μπορούμε παρά να την υποστηρίξουμε. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε πόσο βαριά και ακριβή είναι η σημερινή διαδικασία για να ζητήσει κανείς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ξεχωριστά σε κάθε κράτος μέλος. Εγώ απήχα όμως γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφής ρύθμιση για το γλωσσικό. η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σχέδιο πρότασης δεν ανταποκρίνεται ε, στα αιτήματα των άλλων γλωσσών πλην αγγλικών, γερμανικών και γαλλικών. Και παρακαλώ το ε, αίτημα αυτό να υποβληθεί και στα Ολλανδικά. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν το λόγο έχουν ε, οι συγητές, ε, η επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Μπελέ. Πρόκειται για τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ε, στα τρόφιμα και τις τροφές. Δίνω το λόγο στον κύριο Νικολάζικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η κωδικοποίηση των κανόνων που ισχύουν σίγουρα θα σημάνει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στην νομοθεσία και στα όσα ισχύουν για τη ραδιενέργεια. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η νομική βάση και να την ελέγξουμε. Στη νομική αυτή βάση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι νέες εξουσίες του Κοινοβουλίου σε θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας. Συμφωνώ ότι ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καλή βάση το άρθρο 168 εδάφιο 4β. Πρόκειται για την προστασία της δημόσιας υγείας και για τα ανώτατα όρια για τη μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών. Ευχαριστώ. Συνάδελφος κύριος Ούτζας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις ε, τροποποίησης ε, που κατατέθηκαν με αυτό το κείμενο, το οποίο όμως σε μεγάλο βαθμό δεν κάνει τίποτα άλλο από το να τροποποιεί αυτά τα οποία έχουν ε, ήδη εγκριθεί για τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ραδιενέργειας στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές. Με το περάσει αυτό το ψήφισμα ε, ξεχνάμε τελικά τι, έχει, τι συμβαίνει με τα πυρηνικά κατάλοιπα και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τους κινδύνους που απορρέουν από τα πυρηνικά εργοστάσια. Αυτά εδώ είναι οι συνέπειες ε, που υπάρχουν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, τρόφιμα που έχουν ε, πληγεί και αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Είναι λοιπόν μια διάταξη η οποία απαιτεί την προσοχή μας και εγώ Επί της ουσίας θέλω να πω το εξή. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να υπάρχει μια άμεση ανακοίνωση ε, που ε, θα οδηγεί στο να ε, αποσυρθούν όλα τα επικίνδυνα προϊόντα. Να μην υπάρχει καμία απολύτως εξαίρεση στο, στην υποχρέωση των κυβερνητικών φορέων να αναφέρουν ατυχήματα στην περίπτωση που προκύπτουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Γκζίπ. Ευχαριστώ. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των τροφίμων από επίπεδο ραδιενέργειας ξεκίνησε μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ. Είναι αρκετά δύσκολο και φλέγον ζήτημα το θέμα των πυρηνικών. Η συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί για ενημέρωση και εξυγχρονισμό των τελευταίων ε, των, των διαφόρων διατάξεων. Ε, υπάρχει η διαφυσβήτηση της νομικής βάσης. Εμείς ζητούμε ως νομική βάση το 168, ε, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ κρίνει ως σωστή νομική βάση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η προστασία των κατανολωτών, αλλά ας μην ξεχνάμε και την προστασία των αγροτών, που εξαιτία του πυρηνικού ατυχήματος, ε, καλό θα ήταν να λάβουν κάποια αποζημίωση για τις ε, ζημιές που υπέστησαν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των διαφόρων απειλών. Ε, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ραδιενέργεια μετά από ατύχημα, αλλά και στο περιβάλλον. Ε, ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε εισαγωγή τροφίμων από διάφορες περιοχές του κόσμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να, απαιτούμε αντίστοιχες υψηλές προδιαγραφές ε, και επίπεδα ραδιενέργειας και για τα προϊόντα που εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά θα πρέπει να τηρούν τα αντίστοιχα επίπεδα. Σας ευχαριστώ κύριο Αντωνιώτση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στην πρόταση κωδικοποίησης των τριών κανονισμών που εγκρίθηκαν ε, στις αρχές δεκαετίας του 90 και ορίζουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ραδιενέργειας σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης ε, εδώ έχουμε τη δυνατότητα να εγκρίνουμε ένα κείμενο το οποίο ε, αιτιολογεί την αρμοδιότητα του Συμβουλίου να μπορεί να παρεμβαίνει έτσι ώστε να ληφθούν ταχύτατα τα έκτακτα μέτρα που θα προτείνει η Επιτροπή. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μπελέτ ότι όλα αυτά δεν πρέπει να αποσυνδέονται. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, εφόσον υπάρχουν νέα κριτήρια με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας, να ξεκαθαρίσουμε κατά πόσον αυτό είναι σωστή τροποποίηση για να διατηρηθούν οι αρμοδιότητες ε, τις οποίες, ε, οι οποίες προβλέπονται για το Συμβούλιο και κατά πόσον οι αρμοδιότητες αυτές είναι και σωστά οριζόμενες και περιορισμένες. Πρέπει να προστατεύσουμε τον πολίτη σε περίπτωση ατυχήματος, αυτό αποτελεί και πρέπει να είναι εγγύηση, εξάλλου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η Κομισιόν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα της εποπτείας ε, και να ε, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που εξυπηρετούν το σκοπό. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, διακόπτουμε μέχρι τις 3 η ώρα.